τράπεζες που είναι υπερβολικά μεγάλες ε, για να ε, διασωθούν. Ε, τι γίνεται λοιπόν με την Deutsche Bank, τι γίνεται με τη συγχώνευση αυτή όσον αφορά την χρηματοοικονομική σταθερότητα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Γκίλ. Το λόγο έχει τώρα από το ECR ο κύριος Λούκε για 1,5 λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, έχουμε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα στην Ευρωζώνη, διότι έχουμε ε, τεράστια συσσόρευση μη εξυπηρετούμενων δανείων. 600 δισεκατομμύρια ευρώ, ε, αν όχι περισσότερα, ε, εάν δεν έχουν κρυφτεί, δηλαδή περισσότερα, δεν έχουν καλυφθεί με διάφορα μέτρα Ε, Η πρόταση αυτή δεν λύνει το πρόβλημα, διότι νομοθετικό μέτρο που η νομοθετική πρόταση αυτή δεν ασχολείται με το βασικό πρόβλημα που έχουμε, διότι όλα τα μη εξυπηρετούμενα δανεία, δάνεια που δημιουργήθηκαν ε, στη, κατά τη διάρκεια της κρίσης δεν καλύπτονται από αυτή τη νομοθεσία. Ε, το, η πρόταση αυτή καλύπτει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια από τη στιγμή υιοθέτησή της. Εφόσον λοιπόν τεθεί σε ισχύ το 2019, δεν θα δούμε αμέσως αποτελέσματα, διότι υπάρχει και μία προθεσμία τριών ετών μέχρι τα πρώτα μέτρα ε, διαγραφής. Δηλαδή, μόλις το 2022 θα αρχίσουν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ε, ε, να υπόκεινται στα μέτρα αυτά. Ο όγκος μη εξυπηρετούμενων δανείων που, που θέτει σε κίνδυνο την ε, σταθερότητα των τραπεζών δεν καλύπτεται καθόλου από την πρόταση αυτή. Πολύ συχνά λοιπόν ε, οι πολιτικοί ε, συγχαίρουν τους εαυτούς τους χωρίς καν να έχουν λύσει το πρόβλημα. Πρόκειται για μια τεράστια αποτυχία αυτού του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ κύριε Λούκε. Από το Άλντε ο κύριος Τρεμόσα Ιμπαλσέλς για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε Ντομπρόσκης, καλώς ήρθατε στο Κοινοβούλιο, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν ήταν εύκολο να συμπεριλάβουμε στις προτάσεις μας ιδέες, γιατί οι δύο ε, συντονιστές έκαναν ό,τι μπορούσαν, παρά τις δυσκολίες επειδή μα ενδιαφέρουν πάρα πολύ εκείνοι που επλήγησαν πάρα πολύ λόγω των ε, μη εξυπηρετούμενων δανείων, προσπαθήσαμε λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Είπαμε ότι τα ΜΕΔ είχαν μια εγγενή ανθρώπινη διάσταση. Συσσωρεύονται λόγω κακή εφαρμογή των ε, ευρωπαϊκών νομοθεσιών. Στην αρχή του κανονισμού η Ένωση αναγνωρίζει ότι υπήρχαν σημαντικοί και νομοθεσίε, νομοθετικά κύματα που δεν εφαρμόστηκαν σωστά σε κάποια κράτη-μέλη. Η οδηγία για τι καθυστερημένε πληρωμέ, η οδηγία για του καταναλωτέ και τα ενυπόθηκα δάνεια δεν εφαρμόστηκαν σωστά. Σας προειδοποιώ, αν δεν βελτιώσουμε την ε, εφαρμογή των νομοθεσιών αυτών στα κράτη-μέλη, μπορεί να κινδυνεύσουμε να δούμε ένα νέο κύμα μη εξυπηρετούμενων δανείων σε κάποια κράτη-μέλη τα επόμενα χρόνια, και μπορεί να γίνει και μια νέα τεράστια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση ξανά. Επομένως, σωστή εφαρμογή είναι πολύ σωστή, σημαίνει δέσμευση απέναντι στους κανόνες μας, στις αξίες και στην ένωσή μας. Το Κοινοβούλιο, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να εγκρίνει ένα πακέτο. Χωρίς την οδηγία, ο κανονισμός δεν έχει κανένα νόημα και οι πιστοτικοί οργανισμοί μπορεί να μην έχουν τα νομικά ενάσματα που χρειάζονται, ούτω ώστε να βάλουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην αγορά. Θεωρούμε ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλα, όλο το νομοθετικό πακέτο για τα ΜΕΔ, για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, να εγκριθεί. Είναι δική μα ευθύνη. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Τρεμόσα Ιμπαλσέλ. Από τους πράσινους, ο κύριος Ουρτασούν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η ομάδα μας συμφωνεί με την ανάγκη να μειώσουμε το πακέτο των ΜΕΔ ε, που στους ισολογισμούς είναι πάρα πολύ μεγάλη, όχι μόνο για γιατί λειτουργία ως τροχοπέδι ε, στην οικονομική ανάπτυξη, αλλά και γιατί είναι μια πηγή αβεβαιότητα πάρα πολύ και αστάθεια πολύ σημαντική. Επομένω, ο στόχο είναι πολύ σοβαρό και τον συμμεριζόμαστε. Υπάρχουν όμω δύο κριτήρια τα οποία θα πρέπει να πρετανεύσουν. Το πρώτο είναι να απαιτήσουμε περισσότερες ευθύνε από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όταν δίνουν πιστώσεις. Ε, θα πρέπει να δουν πότε εγκρίνουν αυτές τις πιστώσεις. Και δεύτερον, προστασία του καταναλωτή και ιδίως εκείνων των καταναλωτών που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ε, τις υποχρεώσεις τους γιατί η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων δεν μπορεί να γίνει με το τεράστιο υψηλό κοινωνικό κόστος που έγινε όπως στην περίπτωση της Ισπανίας. Επομένως, Αυτά τα δύο, με αυτά τα δύο στο μυαλό αντιμετωπίσουμε αυτή την συζήτηση. Ε, είδαμε τον καονισμό. ε, δεν μας αρέσει και δεν θα τον ψηφίσουμε. Ε, γιατί? Γιατί οι διατάξεις που μιλούν για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια τα μελλοντικά είναι πολύ χαλαρές. Η Κομισιόν πρότεινε ότι ε, προβλέπονται 8 χρόνια και εσείς προτείνετε μέχρι 9 χρόνια. Εμείς προτείναμε 7 χρόνια. Ε, Επίσης βάζετε, μόνο, λέτε ότι μόνο τρία χρόνια μετά από την έγκρισή του θα μπει σε εφαρμογή αυτός ο κανόνας. Εμείς λοιπόν προτείνουμε αυτός ο κανονισμός να λάβει υπόψη του και τα προηγούμενα μέδα. Από την 1η Μαρτίου δηλαδή, ε, όσα ανοίγματα και δάνεια είναι υπερήμερα, να συμπεριληφθούν και να καλυφθούν. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι και μας ανησυχεί ότι ο κανονισμός και η οδηγία ε, δεν προστατεύουν επαρκώς τον καταναλωτή. Επομένως, ελπίζω ότι κατά τη διαπραγμάτευση οδηγίας θα λάβετε υπόψη σας πολύ περισσότερο τις απόψεις των μικρών πολιτικών ομάδων. Ευχαριστώ, κύριε Ουρτασόν. Από την ΓΚΟΕ, η κυρία Κάθη για ένα μισή λεπτό. Κύριος. Κανένα από τα επιχειρήματα υπέρ της δέσμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν ευσταθούν αν τα εξετάσουμε σοβαρά. Οι υποστηρικτές λένε ότι θα συμβάλλει στην οικονομική σταθερότητα. Αλλά πώς γίνεται η μεταφορά δισεκατομμυρίων ε, κόκκινων δανείων στον μη ρυθμιζόμενο τραπεζικό τομέα να πετύχει κάτι τέτοιο βλέπουμε τελικά ότι η έλλειψη ζήτηση στην οικονομία και η μη χορήγηση πιστώσεων είναι αυτή που περιορίζει τελικά τον δανεισμό. Πρέπει, και είναι σημαντικό μάλλον που ενισχύεται η προστασία του καταναλωτή, αλλά στην ουσία ρίχνουμε τους καταναλωτές ε, ε, στο στόμα του λύκου. Αυτό ακριβώς ε, γίνεται και στην Ιρλανδία ε, που έχει, ε, έχουμε, βλέπουμε πλέον αστέγους και αυτό το φαινόμενο έχει πάρει διαστάσεις άνευ προηγουμένου. Και βλέπω ότι ακολουθείται και μάλιστα ως μοντέλο που, θα, που θέλουμε να εφαρμόσουμε και αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ είναι το ακριβώς αντίθετο, ένα παράδειγμα προς αποφυγή είναι μια ευκαιρία για τις τράπεζες να έχουν τεράστια κέρδη χωρίς ε, κανένα σεβασμό προς ε, τα δικαιώματα των ε, πελατών τους, των οφειλετών που είναι Ευρωπαίοι πολίτες. Δεν μπορούμε να στηρίξουμε αυτή τη δέσμη γιατί δεν θα λύσει το πρόβλημα των κόκκινων δανείων στο δημοσιονομικό μας σύστημα. Απλώς θα περάσει στην γκρίζα οικονομία και θα τους ρίξουμε στα αρπακτικά. ευχαριστώ κύριε Ο Μάρκο Βάλι από το EFTD. Και εγώ και η ομάδα μου είμαστε πολύ ανήσυχοι για τα μέτρα που θα εφαρμοστούν με αυτό το πακέτο για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Γιατί καταρχάς ε, η μελέτη αντικτύπου δεν έγινε. Επομένως, οι επιπτώσεις που θα υπάρχουν στην αγορά κινήτων και η επίπτωση που θα υπάρχει στους καταναλωτές, στις επιχειρήσεις, στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να δούμε ποιες θα είναι. Γιατί το να δίνουμε κίνητρα για την πώληση των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε σύντομο χρονικό διάστημα σε σχέση με μια χρηστή διαχείριση που θα μπορούσαν να κάνουν εσωτερικά οι τράπεζες, αυτό ε, σημαίνει ότι θα υπάρξει κερδοσκοπία. Υπάρχουν διάφορα ταμεία τα οποία ε, έδωσαν και συμβουλές στην ΕΚΤ και θέλουν να βάλουν το χέρι σε, αυτά τα πακέτια, σε αυτό το πακέτο των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Δεν θέλουμε λοιπόν τα σπίτια, τα κίνητα, ε, τα αγαθά των πολιτών να πέσουν στα χέρια των κερδοσκόπων. Ε, και, και μιλάμε για απομείωση του κινδύνου. Ποια είναι η μείωση του κινδύνου για τα παράγωγα ε, που έχουν οι μεγάλε τράπεζε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι θα γίνει με αυτόν τον περίφημο επιμερισμό του κινδύνου. Περιμένουμε ένα πραγματικό επιμερισμό των κινδύνων με το Ευρωπαϊκό Σύστημα των Καταθέσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Βάλλη. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Ζάλστρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή η έκθεση για την ε, κάλυψη ε, ζημιών έχει να κάνει και με την ε, Ένωση Κεφαλαιογορών, όπου υπάρχει μερισμός του κινδύνου. Αλλά στην πρόσφατη έκθεση ε, του Ολλανδικού Φορέα βλέπουμε το συμπέρασμα ότι τελικά ε, αυτός ο κίνδυνος ε, μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση της σταθερότητας και με την ομοιομορφία, την κλίμακα και την συμμετοχή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για τους Ολλανδούς. Αυτό ο οργανισμό είναι αρκετά γνωστό ίδρυμα. Επομένω, φαντάζομαι ότι και οι συγητέ το έχουν λάβει υπόψη. Επομένω, Πρόεδρε, παραμένει μόνο το ερώτημα γιατί ε, επιθυμούν ε, να ακολουθήσουν αυτή την άγουσα οι συγητές. Ευχαριστώ. Ο κ. Φουντούλης. Προσεγγίζει το σοβαρό αυτό ζήτημα κυρίως από τη σκοπιά των τραπεζών και όχι με γνώμονα την προστασία των καταναλωτών. οι τράπεζες αποτελούν σημαντικό πυλώνα της οικονομίας των κρατών μελών. πιθανή κατάρρευσή τους στη δεδομένη χρονική στιγμή θα σήμαινε τρομακτικές δυσκολίες για την καθημερινότητα των πολιτών αλλά και για τα ίδια τα κράτη. πρέπει να εντοπιστούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές και να υποχρεωθούν να πληρώσουν. οι τράπεζες όμως ευθύνονται για την ανεξέλεγκτη χορήγηση δανείων χωρίς εγγυήσεις εκατομμύρια πολίτε στα κράτη μέλη τη ενώσεω εξαιτία κυρίω τη οικονομική κρίση δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα χρέη του και κινδυνεύουν να χάσουν ακόμα και την κατοικία του. οι τράπεζε μέσω των ανακεφαλαιοποιήσεων από χρήματα των πολιτών συνεχίζουν να λειτουργούν. για του πολίτε που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωση λόγω των χρεών του θα πρέπει να ληφθούν μέτρα όπω προστασία τη κύρια κατοικία του και παροχή ευκολιών στην αποπληρωμή των δανείων του ειδικά για του άνεργου χαμηλόμισθου και τι πιο ευάλωτε κοινωνικέ ομάδε. ευχαριστώ. Sorry. There was no translation. Can you ask if the translation is okay? Ah. Uh, is there a problem with interpretation? Υπήρξε πρόβλημα με τη διερμηνία. Uh, kein Deutsch, oder? Okay. Δεν ακούστηκαν τα γερμανικά. Um, what can we do? you Just continue. Yeah. Okay. I think we've solved the problem, I hope. Νομίζω λύθηκε το πρόβλημα, ελπίζω τουλάχιστον. Παρακαλώ συνεχίστε λοιπόν. So, colleague, you can continue. Συνάδελφε, μπορείτε να προχωρήσετε, να συνεχίσετε. Okay. Right. Okay. Um, hyvä, teille. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Μαυρίδη. Δύο λεπτά παρακαλώ. Πολύ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα για το οποίο αυτό το κείμενο αποτελεί ένα βήμα επιπλέον μπροστά. επιδίωξη είναι η μείωση με ένα αποτελεσματικό τρόπο των μη εξυπηρετούμενων δανείων και ταυτοχρόνως χωρίς να δημιουργούνται αρνητικές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία και στους δανειολήπτες. ως εδώ όλα καλά. τρία σημεία. πρώτον η προστασία των δανειοληπτών με δεδομένο ότι η τράπεζα είναι εκ των πραγμάτων ο δυνατός και ο δανειολήπτης καταναλωτής είναι εκ των πραγμάτων ο αδύνατος όπως καθορίζεται και στη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή οδηγία περί καταχρηστικών ρητρών σημαίνει ότι εμείς θα πρέπει να παρεμβαίνουμε και ιδιαίτερα η ευρωπαϊκή επιτροπή να διερευνά καταγγελίες για μη αποτελεσματική εφαρμογή της συγκεκριμένης οδηγίας σας αναφέρω λοιπόν ότι στην περίπτωση ιδιαίτερα της κύπρου η ευρωπαϊκή οδηγία η συγκεκριμένη δεν εφαρμόζεται με αποτελεσματικό τρόπο και σε άλλα κράτη μέλη δεν εφαρμόζεται με ομοιόμορφο τρόπο. το δεύτερο σημείο risk sharing. εδώ θα επαναλάβω κάτι που είπε συνάδελφός μου ιδεολογικοί λόγοι αλλά και θα προσθέσω ειδικά συμφέροντα κάποιων κρατών μελών εμποδίζουν την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής τραπεζικής ένωσης με τον τρίτο πυλώνα που ήταν και παραμένει το ζητούμενο πανευρωπαϊκή εγγύηση των καταθέσεων. χωρίς αυτό δεν μπορούμε να μιλούμε για ουσιαστικό ανταγωνισμό ο οποίος να είναι δίκαιος ανάμεσα στις τράπεζες των κρατών μελών. και το τρίτο σημείο, πρόσφατα στην κύπρο είχαμε ένα πόρισμα από την ερευνητική επιτροπή που διορίστηκε σε σχέση με την κατάρρευση της συνεργατικής τράπεζας. το πρόβλημα ήταν εξ αρχής όπως διαφάνηκε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. σας ομολογώ όμως ότι το πόρισμα καταλήγει σε κάτι που αφορά τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. εξαπατήθηκαν από τις συγκεκριμένες αρχές της κυβέρνησης στην κύπρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μαυρίδη, προχωράμε στον επόμενο μιλητή, τον κύριο Ζόγκ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκαναν πρόοδο σε ό,τι αφορά την ποιότητα του χαρτοφυλακίου τους και σε ό,τι αφορά τον όγκο των μη εξυπηρετούμενων δανείων για να μην υπάρξει τέτοια συσσόρευση στο μέλλον, θα πρέπει να εισαχθούν επιπλέον μέτρα. Γι' αυτό ακριβώς η Πολωνία είναι ικανοποιημένη για αυτή την νομοθετική πρόταση. Θα ήθελα όμως να σε πιστήσω την προσοχή σε δύο θέματα. Καταρχήν, αυτή η καθολική προσέγγιση που έχουμε εισαγάγει σήμερα δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των κρατών μελών παραδείγματο χάρη των διαδικασιών που έχουν σε εθνικό επίπεδο. Δεύτερον, θα πρέπει να κάνουμε μία μελέτη αντικτύπου. Θα πρέπει να δούμε σε ποιο βαθμό αυτό θα επηρεάσει την κατάσταση των επιχειρήσεων, των οικοκυριών και την οικονομία των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριο Ζούγκ. Ο κύριος Παπαδημούλης έχει το λόγο ασφαλώς πρέπει να μειώσουμε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια γιατί είναι πάρα πολύ ψηλά 600 δισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά πρέπει να το κάνουμε εξασφαλίζοντας μια επαρκή προστασία των καταναλωτών απέναντι σε κερδοσκοπικές πρακτικές. Και αυτό δεν το κάνει ούτε η πρόταση της Κομισιόν με επάρκεια, ούτε η κοινή πρόταση συμβιβασμού ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και την Σοσιαλιστική Ομάδα. Και επίσης αν θέλουμε ένα υγιές τραπεζικό σύστημα πρέπει να εξασφαλίσουμε και ότι ο μη ρυθμιζόμενος τραπεζικός τομέας θα υπάγεται και θα υπακούει στους ίδιους κανόνες διαφάνειας και λογοδοσίας και αυτό πάλι δεν εξασφαλίζεται με αυτή την πρόταση. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να το στηρίξουμε. Και επιπλέον είμαστε αντίθετοι με τη σαλαμοποίηση του προβλήματος και με τις διαρκείς αναβολές. Κυρία Εστέρ Ντελάγκετ, έχετε επί τέσσερα χρόνια το φάκελο του ίντις στα χέρια σας και κρατάτε καθυστέρηση και δεν έχει γίνει τίποτα και τελειώνει η θητεία. Έχει μειωθεί ο κίνδυνος αλλά το risk sharing, ο επιμερισμός του κινδύνου δεν έχει προχωρήσει ένα βήμα. Ενώ το προτείνει η Κομισιόν, το υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ένα μεγάλο τμήμα του Ευρωκοινοβουλίου. Έτσι, με τη σαλαμοποίηση δεν θα πετύχουμε τίποτα και ο κανονισμός δεν έχει κανένα νόημα χωρίς την παράλληλη οδηγία. πολύ λίγα πολύ αργά αυτά που έχετε προτείνει και γι' αυτό δεν μπορούμε να τα στηρίξουμε. Ευχαριστούμε κύριε Παπαδημούλη. Ο κύριος Αριανόπουλος. Ένα λεπτό. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αφού χάρισε 20 εκατομμύρια προχθές στους φαρμακοβιομήχανους συμφώνησε σε εθελοντική όχι υποχρεωτική φορολόγηση με ψίχουλα των εφοπλιστών φοροαπαλλάσσει τράπεζες και φαντς επί ετία, βγάζει τώρα τα σπασμένα στις πλάτες του λαού καταργεί πλήρως την όποια δικαστική προστασία της πρώτης κατοικίας χιλιάδων λαϊκών οικογενειών από πληστηριασμούς. το 19 προγραμματίζονται 20.000 πληστηριασμοί με μόνη απόφαση των τραπεζών και των φαντς όπου μεταβιβάζονται χιλιάδες δάνεια και τραπεζοϊπάλληλοι που τους περιμένει η απόλυση λεόντιες ρυθμίσεις δανείων για ένα μόνο χρόνο που είναι αδύνατο να τηρηθούν για τους ελάχιστους που θα μπουν σε αυτές λόγω αυστηρότατων κριτηρίων. ελεύθεροι πληστηριασμοί για τα κόκκινα δάνεια από εδώ και πέρα. οι συζητήσεις συριζα eurogroup δεν αλλάζουν τη συναπόφασή τους για εκατό χιλιάδες πληστηριασμούς σε μια τριετία. Και άλλη δηλαδή ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών για να χρηματοδοτήσουν το κεφάλαιο. μνημόνιο και εποπτεία διαρκείας. κανένα ψευτοπροοδευτικό μέτωπο δεν κρύβει αυτή τη βαθιά αντιδραστική πολιτική. άλλωστε και εδώ μέσα η χρυσή αυγή προέβαλε πρώτα απ' όλα τη διάσωση των τραπεζών και όχι των δανειοληπτών. το σύνθημα κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη να κινητοποιήσει τις εργατικές λαϊκές οικογένειες να γίνει κριτήριο στάσης τους στις εκλογές. ευχαριστώ κύριε Ζαριανόπουλε. Φρουντζούλικα, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Συνάδελφοι, Επίτροπε, η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για να αντιμετωπίσουμε τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για να γίνει πιο ανθεκτικό το, οικονομικό σύστημα, το χρηματοοικονομικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα αυτό είναι κυρίως αρμοδιότητα των ε, ε, τραπεζών και των κρατών μελών. Υπάρχει ενωσιακή διάσταση στην μείωση του μεγάλου όγκου των ε, μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και η αποτροπή της ισόρευσής τους στο μέλλον. Έτσι μπορούμε να προλάβουμε συστημικούς κινδύνους. Πιστεύουμε ότι έτσι θα μπορέσουμε να προλάβουμε κλειδονισμούς ε, και να έχουμε επιμερισμό των κινδύνων. Η πρόταση αυτή είναι απαραίτητη διότι στόχο έχει την ε, πρόληψη των ε, μεγάλων απολειών στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Φροντζούλικα. Ο κύριος Πακέτα, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. 714 δις ευρώ. Αυτό το τεράστιο ε, ποσό λοιπόν ε, είναι κάτι το οποίο 10 χρόνια μετά την χρηματοπιστική κρίση εξακολουθεί να παραμένει στους ισολογισμούς των ευρωπαϊκών τραπεζών και αυτό έχει συνέπειες. Στην Ιταλία, όπου τα κόκκινα δάνεια είναι τεράστιο πρόβλημα, η Ιταλική κυβέρνηση τον Ιανουάριο ε, βοήθησε την τράπεζα Καρίγκια και έτσι θεωρώ ότι είναι, ε, έχει έρθει η ώρα να υιοθετήσουμε ε, μέτρα και μάλιστα έχουμε καθυστερήσει και θα πρέπει να πάμε περισσότερο, παραπέρα. Αλλά οι μακρόν αυτή τη Ευρώπη συνεχώ ε, θέλουν να συζητάνε άλλα πράγματα. Αλλά αν ε, ξεκινούσαμε από ο καθένα τα δικά του, και αν ρύθμιζε ο καθένα τα δικά του, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος Λιμπεράτσκι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, πράγματι σήμερα εξετάζουμε ένα πρόβλημα το οποίο είναι πραγματικά ε, πονοκέφαλος και για τις τράπεζες και για τους πολίτες. Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι ιδιαίτερα πιστικό αυτό το κείμενο. Έχουμε εργαστεί επί μακρόν, αλλά πρόκειται για ένα πολύ σύνθετο ζήτημα. Το πιο σημαντικό είναι ο επιμερισμός του κινδύνου μεταξύ των τραπεζών και των οφειλετών. Και πρέπει εδώ να έχουμε κατά νου ότι υπάρχουν και διαφορετικές κατηγορίες ε, οφειλετών και διαφορετικές κατηγορίες επιστώσεων. Έχουμε καταναλωτικά, επενδυτικά δάνεια κτλ. Πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα καλό σύστημα, το οποίο ε, θα αποτρέπει την ε, δημιουργία ε, μη εξυπηρετούμενων δανείων. Αυτά που έχουμε προβλέψει τώρα είναι επαρκή. Πρέπει να προστατεύσουμε τι τράπεζε, αλλά παράλληλα να προστατεύσουμε και του επενδυτές και του καταναλωτέ, και αυτό δεν είναι εύκολο. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κ. μαριά. Μιλούμε για τα κόκκινα δάνεια στην Ένωση, τη στιγμή που στην Ελλάδα οι φτωχοποιημένοι από τα μνημόνια Έλληνε, κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια του από τα κοράκια. Παρά ότι ο ελληνικό λαός με την υπερχρέωσή του λόγω μνημονίων έσωσε του ξένου δανειστέ, αλλά και τι τράπεζε παρότι η ελλάδα χρεώθηκε με διακόσια δισεκατομμύρια ευρώ τελικά η τρόικα με επικεφαλή στην εκτ και τον ντράγκη απαιτούν από τις τράπεζες το ξεπούλημα των κόκκινων δανείων στα κοράκια αντί πινακίου φακής. η κυβέρνηση τσίπρα αλλά και οι προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις άφησαν το πρόβλημα των κόκκινων δανείων να διωγγωθεί. τώρα η κυβέρνηση τσίπρα καταργεί την προστασία πρώτης κατοικίας και ρίχνει τους δανειολήπτες βορρά στους τοκογλύφους. μόνη λύση η δημιουργία ταμείου σωτηρίας δανειοληπτών με κρατική παρέμβαση που θα αγοράσει τα κόκκινα δάνεια στην τιμή πρώτης προσφοράς που κάνουν τα κοράκια. Πρόταση που υποβάλαμε εδώ και δύο χρόνια. Στοπ εδώ και τώρα στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Αυτό πρέπει να είναι το κεντρικό σύνθημα και στις επικείμενες ευρωεκλογές. Γιατί για την Ελλάδα υπάρχει άλλος δρόμος. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαριά. Έχουν ζητήσει και άλλοι συνάδελφοι το λόγο. Δίδικα σε Catch the Δύο συγκεκριμένα. Ο κύριος Τραγιαυσκή. Είτε είναι 600 είτε 700 τα δις των ε, μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Αλλά δεν είναι τόσο επώδυνο σήμερα, καθώς η οικονομική ανάπτυξη αυξάνεται. Είναι πολύ πιο δύσκολο και ε, επώδυνο αυτό το πρόβλημα σε περίοδους ε, στασιμότητας αλλά δεν έχουμε καταδείξει ακόμα τις αιτίε του προβλήματος. Είναι το σύστημα, είναι τα λάθη των τραπεζών. Πρόκειται για συγκεκριμένες ενέργειες, συγκεκριμένων οντοτήτων, φορέων ή προσώπων. Εγώ, για παράδειγμα, στην Επιτροπή Κατά της Τρομοκρατίας ασχολούμαι με τα bitcoin και έχω εξετάσει και τις τραπεζικές δραστηριότητες και θεωρώ ότι μέχρι το τέλος της θητείας θα πρέπει να εισαγάγουμε διατάξεις δεσμευτικές. Καλό είναι που έχουμε αυτή την έκθεση, αλλά πρέπει να πάμε παραπέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τέλος, ο κύριος Επιτίδιος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε ε, οι τράπεζες ε, αποτελούν ε, τμήμα της οικονομίας ενός κράτους. είναι λοιπόν λογικό να επιδεικνύεται ενδιαφέρον ώστε να επιβιώσουν να μην καταρρεύσουν και να μπορέσουν να χορηγήσουν δάνεια τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την εξέβρεση εργασίας και απασχολήσεως. πρώτιστος όμως αντικειμενικός σκοπός δεν είναι η επιβίωση των τραπεζών αλλά είναι η βοήθεια των δανειοληπτών οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν τα δάνεια τα οποία έχουν λάβει λόγω της οικονομικής κρίσεως ο αριθμός αυτών των ανθρώπων είναι πολύ μεγάλος σε όλα τα κράτη της ευρωπαϊκής ενώσεως. τραγικές διαστάσεις λαμβάνει αυτό το φαινόμενο στην ελλάδα όπου εκατομμύρια έλληνες λόγω της οικονομικής καταστροφής της χώρας εξαιτίας των μνημονίων δεν έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν τα δάνειά τους τα οποία γίνονται κόκκινα και καθημερινά χιλιάδες από αυτούς χάνουν τα σπίτια τους. πρόσφατα πριν δύο ημέρες ένας άνδρας 54 ετών αυτοκτόνησε όταν οι κρατικοί υπάλληλοι ήρθαν να κατασχέσουν το σπίτι του. Αυτή πρέπει να είναι η προσπάθεια που οφείλουμε να καταβάλουμε. Να προστατεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους, να προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να αποπληρώσουν τα δάνεια τα οποία έχουν λάβει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επιτίδια. Τώρα θα ακούσουμε τον Επίτροπο, τον κύριο Ντομπρόφσκης. Παρακαλώ. Uh, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές, ε, κυρίες και ε, κύριοι συγητές. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την δουλειά που έχετε κάνει και τους σκιώδεις εισηγητές για τις επιτυχείς διαπραγματεύσεις πάνω στο θέμα αυτό. Θα ήθελα να τονίσω ότι αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία δείχνει ότι η Ένωση είναι πράγματι ενωμένη και μπορεί να αναλάβει αποφασιστική δράση για να ενισχύσει και να σταθεροποιήσει τον τραπεζικό τομέα, να τον κάνει ανθοκτικό σε μελλοντικού κλειδονισμούς και να τον κάνει ικανό να δανείζει χρήματα στην πραγματική οικονομία. Αυτό είναι σημαντικό για τη μελλοντική μας ευημερία και μια ανθεκτική οικονομική και νομισματική ένωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Ευχαριστούμε, Πίτροπε. Και τώρα θα ακούσουμε τους εισηγητές κυρία Ντελάγκη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δύο ακόμα παρατηρήσεις. Γιατί ακούστηκαν πολλά σχόλια για ε, το σύστημα εγγύηση καταθέσεων. Πρέπει να, πάρουμε, να κάνουμε ένα βήμα προ τα πίσω και να θυμηθούμε ότι στις περιόδους, ε, την περίοδο τη κρίση ζητήσαμε πολλά από του ε, Ευρωπαίου φορολογούμενου ό,τι αφορά την εξασφάλιση και τη διάσωση τραπεζών και κρατών μελών αλλά έχουμε πει ότι ω εδώ, την, την επόμενη φορά που θα χρειαστεί μια διάσωση μια τράπεζα, θα είναι ο φορολογούμενο, αλλά ο μέτοχο που θα λάβει τον ε, λογαριασμό. Είδαμε ότι σε κάποιε χώρε. Και πάλι όμως ε, το κράτος ε, τίθεται εγγυητής για την διάσωση μιας τράπεζας και γι' αυτό θεωρώ ότι όταν υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές μεταξύ κρατών μελών σε ό,τι αφορά την χρήση δημοσίου χρήματο για την διάσωση του κράτου της τράπεζας, ε, και πάλι βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ενότητα για έναν ανιαίο καθεστώ ε, εγγύηση καταθέσεων στην Ευρώπη. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Υπάρχει μια καλή πρόταση να ξεκινήσουμε με την υποχρεωτική στήριξη ρευστότητας. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι κάποιες πολιτικές ομάδες θέλουν από τώρα ε, την εγγύηση ότι θα πάμε σε ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο. Και, και η πρόσφατη διάσωση τραπεζών στην Ιταλία και το γεγονό ότι κάποιε πολιτικέ ομάδε είναι κατά ε, τη σημερινή νομοθεσία για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μα δείχνουν ότι ακόμα δεν υπάρχει η πολιτική στήριξη δεν υπάρχουν κράτη-μέλη που ακόμα δεν μπορούν να λάβουν την υπεύθυνη στάση που απαιτείται. Δεύτερον, προς τον συνάδελφο Ζάλιστρα, που ακολούθησε λίγο το πρότυπο Φαράτζ, που ήρθε για δύο λεπτά, έκανε την παρέμβασή του, έφυγε. Ε, θεωρεί ότι δεν είναι αρκετά ισχυρή ε, αυτή η πρόταση. Όμω, σε αυτές τις διαπραγματεύσεις τον εκπροσώπησε άλλο συνάδελφο από την Ιταλία της δική του πολιτική ομάδας που ανέφερε ότι θα πρέπει σε αυτή την πρόταση να έχουμε ε, πολύ μακρι... Ε, πιο μακροπρόθεσμους ε, στόχους. Και 20, χρόνια, συγγνώμη, 20 ώρες είχαμε διαπραγματεύσεις με τους συναδέλφους. Το κόμμα του κυρίου Ζέλστρα, το PVV, δεν, δεν συμμετείχε καθόλου. Επομένω, τελικά η συμβολή του κυρίου Ζέλστρα ήταν μηδενική, ούτε καν mail δεν μου έστειλε. Επομένω, να πω προς τον PVV, είτε θα κάνετε τη δουλειά σας ε, και θα μου στείλετε ένα mail ή θα συμμετάσχετε στη συζήτηση, είτε θα σοπάσετε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ντελάνε. Ο κύριος Γκουαλτιέρη, παρακαλώ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ πιστεύω ότι σε αυτή τη συζήτηση φάνηκε ότι εγκρίναμε ένα ισορροπημένο κείμενο, ότι ακούσαμε λιγάκι κάποια σλόγγαν και προπαγάνδα ένθεν και ένθεν, ε, ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Και στον κύριο Βάλλη θα ήθελα να πω ότι ε, πρέπει να δείξουμε λίγη σοβαρότητα. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι είναι ένα κείμενο το οποίο μαλάκωσε την πρόταση της Κομισιόν, είναι πιο ισορροπημένο. Το να μας κατηγορείτε λοιπόν ότι φτιάξαμε ένα πολύ σκληρό και προπαγανδιστικό κείμενο είναι λάθος. Είναι απλώς προπαγάνδα. Επίσης, συμφωνώ με την κυρία Τερλάγκεν ότι όλους αυτούς τους συναδέλφους δεν τους είδαμε καθόλου. Δεν παρενέβησαν. Ε, όλοι αυτοί που μας λένε ότι έπρεπε να ήμασταν πιο σκληροί στις διαπραγματεύσεις, και μας κατηγορούν ότι δείξαμε μεγάλη χαλαρότητα, ας πούμε. Στην πραγματικότητα, εμείς αναλάβαμε τις ευθύνες μας, αντιμετωπίσαμε ένα πολύ λεπτό και δύσκολο θέμα, καταφέραμε να φτιάξουμε ένα καλό κείμενο σε πολύ μικροχρονικό διάστημα και αυτοί απουσίαζαν. Και αυτό δείχνει όμως την ικανότητα του Κοινοβουλίου να παράγει νομοθεσία και όταν δεν λειτουργεί κάτι καλά, κάποια αρχή, κάποιος φορέας δεν τα πάει καλά, και όταν χρειάζονται λύσεις ε, για προβλήματα στην πραγματική οικονομία, το Κοινοβούλιο διορθώνει τα προβλήματα και εξασφαλίζει την απαραίτητη τη, τη μείωση του κινδύνου λόγω των μη εξυπηρετούμενων δανείων για το καλό των οφειλετών, των πολιτών, των καταναλωτών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και παράγουμε ένα, με αυτόν τον τρόπο μια νομοθεσία, ένα καονισμό δηλαδή που θα έχει σημαντική επίπτωση γιατί θα υπάρχει μεγαλύτερη σύνεση, δεν θα υπάρχουν πλέον κακές πρακτικές που θα οδηγούν σε υπερβολική συσσόρευση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και θα είναι όλα πιο διαχειρίσιμα χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία. Ευχαριστώ λοιπόν την κυρία Ντελάγκη, ευχαριστώ την Κομισιόν και όλους τους συναδέλφους που στήριξαν τη δουλειά μας, καθώς και το Συμβούλιο που μας επέτρεψε να συζητήσουμε στα πλαίσια του τριμερού διαλόγου σε χρόνο ρεκόρ, ίσως τον πιο σύντομο τριμερή διάλογο κάναμε, γι' αυτό τα καταφέραμε να βάλουμε αυτόν τον κανόνα στην επίσημη εφημερίδα σε χρόνο ρεκόρ. Όλα αυτά σε χρόνο ρεκόρ. Ευχαριστώ. Ε, ε, Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκουαλτιέρη. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση και αύριο θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία. Φτάνουμε έτσι στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Προσωρινή έκθεση των συναδέλφων Περέιρα και Μάνκα για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου. Το λόγο δίνω πρώτα στους δύο εισηγητές. Πρώτα στον κύριο ε, Περέιρα, τέσσερα λεπτά. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ επίτροπε, η μεταρρύθμιση του μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ε, είναι πολύ σημαντική γιατί είναι μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση. Είναι μια απαραίτητη διαδικασία για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες ελλείψεις στην αρχιτεκτονική του ευρώ που αποκάλυψε με δραματικό τρόπο η χρηματοπιστωτική κρίση. Αυτή την έκθεση το Κοινοβούλιο συμμετέχει με πολύ σημαντικό ρόλο στην διαδικασία αυτή. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή μου, τον κύριο Μάνκα, για την θαυμάσια συνεργασία που είχαμε τους τελευταίους μήνες. Ευχαριστώ επίσης ε, και τους σκιώδεις συζητητές από τις διάφορες πολιτικές ομάδες για το πνεύμα αυτό συνεργασίας που επέδειξαν, που μας επέτρεψαν να καταλήξουμε σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Με αυτή την έκθεση το Κοινοβούλιο ε, διαμορφώνει μια στρατηγική σε δύο χρόνους για το μεσοπρόθεσμο και το μακροπρόθεσμο χρονικό διάστημα βλέπουμε ποια είναι το δικό μας όραμα, ούτω ώστε να έχουμε ένα ευρωπαϊκό μηχανισμό σταθερότητας για να καταστεί και αυτός ο μηχανισμός ένα πραγματικό θεσμικό όργανο ε, με διακυβέρνηση και σοβαρή και υπό τον δημοκρατικό έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν θα μπορέσει να γίνει βεβαίως αυτό εν μία νυχτή. Βραχυπρόθεσμα λοιπόν υπερασπιζόμαστε την πρόοδο στη μεταρρύθμιση του συστήματος σταθερότητας με την ε, ε μεταρρύθμιση της διακυβερνητικής συνθήκης από τις οποίες απορρέπτει, απορρεί, απορρέει. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε ακόμα για το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, γιατί θα μπορούσαν να δημιουργηθούν προβλήματα όσον αφορά τις αρμοδιότητες για την νομισματική πολιτική. Ε, η αρμοδιότητα της νομισματικής πολιτικής αφορά την ΕΚΤ πάντα. Υπάρχουν και άλλα σημαντικά στοιχεία που πρέπει να μας απασχολούν. Θα πρέπει να υπάρξει δημοκρατικός έλεγχος του μηχανισμού ε, και αυτός να είναι στα χέρια του Κοινοβουλίου. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων για να ενισχύσουμε το διάλογο για να ενισχύσουμε την ε, κοινοβουλευτική εξέταση και έλεγχο και θα πάμε και πιο μακριά. Προτείνουμε ο Διευθυντή του Μηχανισμού Σταθερότητα να εκλέγεται εδώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εν συνεχεία, προβλέπουμε την ενίσχυση του ρόλου του μηχανισμού για να προωθήσουμε την χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Για την απάντηση στα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά σοκ με την αναθεώρηση των αρμοδιοτήτων του, λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως τη, τις αρμοδιότητες για τη μακροοικονομική εποπτεία που είναι καθήκον και αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τέλος, θα πρέπει να έχουμε μια μεγαλύτερη αυτονομία ε, σε σχέση με το του. Θα πρέπει να δώσουμε στο μηχανισμό αρμοδιότητες ούτως ώστε αυτό το ενιαίο ταμείο να είναι λειτουργικό, για να, το Ταμείο Εξυγίασης δηλαδή, ε, να λειτουργήσει καλά για να μας επιτρέψει την Τραπεζική Ένωση. Θα πρέπει να υπάρχει βεβαίω και το δημοσιονομικό υπόβαθρο. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού ε, Μηχανισμού Σταθερότητας, που είναι σημαντική φάση της όλης διαδικασίας. Ελπίζω λοιπόν το Συμβούλιο να ακούσει τις προτάσεις και τις υποδείξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ούτω ώστε να προχωρήσουμε όλοι μαζί προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστώ κύριε Περέιρα. Περνάμε στον δεύτερο εισηγητή, τον κύριο Μάνκα. Τέσσερα λεπτά έχετε στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνάδελφοι. Θα θυμούνται όλοι την οικονομική βοήθεια προς την Ελλάδα, τη χώρα που υπέφερε περισσότερο από την ε, χρηματοπιστωτική κρίση. Τότε οι χώρες της Ευρωζώνης δημιούργησαν ε, τον Ευρωπαϊκό ε, Μηχανισμό Σταθερότητας που ήταν προσωρινός αρχικά, αργότερα έγινε μόνιμος ε, και είχαμε και τα ευρωομόλογα. Είδαμε λοιπόν ε, χώρες όπως είναι η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ελλάδα ε, και η Κύπρος να χάνουν την πρόσβασή τους στις αγορές. Οι χώρες αυτές έπρεπε να εφαρμόσουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, μέτρα δηλαδή για να γίνουν πιο ισχυρές οι οικονομίες τους και να αποτρέψουν ζημίες όχι μόνο στην Ευρωζώνη αλλά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας κοιτάξουμε λοιπόν τις χώρες αυτές. Ε, χάρη στην Ευρωπαϊκή Συνεργασία η Ιρλανδία έχει τους ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ε, Ισπανία έχει σπάσει τα ρεκόρ, τα το ιστορικό της ρεκόρ όσον αφορά ε, την, τις εξαγωγές. Ε, η Κύπρος πηγαίνει πολύ καλύτερα και η Ελλάς πια μπορεί να βρίσκει χρηματοδότηση στις διεθνείς αγορές. Έχουν δημιουργηθεί ε, εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις απασχόλησης και σημειώνεται σημαντική οικονομική ανάπτυξη. Πριν λίγες μέρες η Moody's ε, ε, βελτίωσε την ε, βαθμολογία της Ελλάδας σε κατά δύο βαθμίσεις στο Β1 και διαπιστώνεται ότι έχουν εφαρμοστεί ήδη μεταρρυθμίσεις και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για περαιτέρω ανάπτυξη και πολύ χαμηλός κίνδυνος επαναφοράς στην προηγούμενη κατάσταση. Στην Σλοβακία ε, έπεσε η κυβέρνησή μας ε, το 2012, χάρη όμως ε, στην ευρωπαϊκή συνεργασία. Το ευρώ είναι πολύ πιο ανθεκτικό στις κρίσεις και η υποστήριξη για το ευρώ βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα από τη δημιουργία του. Μετά τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας είδαμε ότι ε, ο διακυβερνητικός ε, χαρακτήρας μειώνει τη δυνατότητα ανταπόκρισης σε οικονομικούς κλειδονισμούς. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας του. Είναι απαραίτητο το μελλοντικό πλαίσιο να αντικατοπτρίζει και τις θέσεις των Εθνικών Κοινοβουλίων. Όταν μιλάμε για τους μελλοντικούς πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, θα πρέπει το Κοινοβούλιο να συμμετέχει στην διαδικασία απαλλαγή και να ελέγχει όλες τις πτυχές ε, της διαδικασίας του προϋπολογισμού, όπως άλλωστε και ε, το ελεγκτικό συνέδριο. Οι οικονομικοί πόροι και ε, τα εργαλεία της μεταρρύθμισης ε, θα πρέπει να επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να έχουν ε, χρηματοοικονομική βοήθεια προτού να αντιμετωπίσουν ε, σημαντικές δυσκολίες στην αναζήτηση χρηματοδότησης στις διεθνείς αγορές. Και μπορούν τα μέτρα να συμπληρωθούν από μέτρα του προϋπολογισμού για να έχουμε σταθεροποίηση των επενδύσεων και σύγκληση οικονομική προς τα πάνω. Επίσης, ο μηχανισμός αυτός δεν θα πρέπει να είναι ανοιχτό μόνο στι χώρες ε, της Ευρωζώνης, αλλά σε όλα τα κράτη-μέλη. Αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω ότι η κοινή μα αυτή προσπάθεια θα οδηγήσει σε περισσότερη ασφάλεια και βεβαιότητα όχι μόνο για την Ευρωζώνη, αλλά για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. ευχαριστώ. τον κύριο Μάνκα. Ο λόγος τώρα στον ε, Επίτροπο. Κύριε Ντομπρόφσκης, έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεχώς ε, διαδραματίζει πρωτοποριακό ρόλο στη συζήτηση ε, για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση και έχει δείξει και μεγάλη στήριξη στην πρωτοβουλία της Κομισιόν για την ενίσχυση της ε, δομής της Ευρωζώνης. Και η σημερινή συζήτηση για την ενδιάμεση πρόταση, πρόταση ενδιάμεσης έκθεσης της Κομισιόν είναι ένα ακόμα βήμα προ αυτήν την κατεύθυνση. Εξ ονόματο τη Επιτροπή, θα ήθελα και να ευχαριστήσω όσου σχολίασαν και του συζητητέ ιδιαίτερω, κ. Σιλβία Περέιρα και Μάνκα, και του σκιώδει συζητητέ για τα όσα έχουν κάνει για αυτό το φάκελο. Επί ευκαιρία, θα ήθελα να ευχαριστήσω και όσου συνεργάστηκαν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία χρόνια για την ολοκλήρωση τη Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Η Κομισιόν χαιρετίζει την ενδιάμεση έκθεση και συμφωνεί με τα πιο σημαντικά μηνύματα σε έδρε γραμμέ. Πιο συγκεκριμένα, στηρίζουμε το Κοινοβούλιο στην προσπάθεια ενσωμάτωση ε, του μηχανισμού σταθερότητα στο ενωσιακό πλαίσιο αυτό όπως ξέρετε ήταν και πρόταση, στόχος της δικής μας πρότασης από το φθινόπωρο του 2012. Ο ESM έχει αποδείξει ε, την ε, δυνατότητά του να, διασφαλίζει, να συμβάλλει στη διασφάλιση της σταθερότητας στην Ευρώπη. Και η ενσωμάτωσή του στο ενωσιακό πλαίσιο ε, θα ενισχύσει αυτό το ρόλο, αλλά και τη λογοδοσία και δημοκρατικότητα και διαφανή λειτουργία αυτού του μηχανισμού, κάτι το οποίο έχετε εξετάσει και εσείς ε, στην έκθεσή σας. Ένα άλλο σημαντικό σημείο που αναφέρετε και με το οποίο συμφωνούμε είναι η αναγκαιότητα ε, τήρησης των κοινών κανόνων ε, διακυβέρνησης από όλα τα κράτη-μέλη για να μην υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις ή άλλες επιρροές προς τα κράτη-μέλη και τα χρηματοπιστωτικά του ιδρύματα και να υπάρχει πλήρη συμμόρφωση με τον ουσιακό δίκαιο. Χαιρετίζω και την έκκλησή σα ε, για ε, εισαγωγή του κοινού μηχανισμού ασφαλείας ε, μέχρι το 2020. Τέλος, για την ονομασία. Εμείς προτείναμε το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, γιατί αυτή ήταν η κοινή ορολογία τη συζήτηση πολιτική. Όμω σημειώσαμε τι επιφυλάξει και αντιρρήσει και τη ΕΚΤ και του Κοινοβουλίου και είμαστε διατεθειμένοι να το επανεξετάσουμε. Θα μπορούσαμε να το διατηρήσουμε με τη σημερινή του ονομασία Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα. Υπάρχουν νέες εξελίξεις βέβαια. Ε, πιο συγκεκριμένα κάποια κράτη-μέλη αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αναθεώρηση της ε, συνθήκης ESM στο διακυβερνητικό πλαίσιο. Συνεχίζονται αυτές οι διεργασίες και θέλουμε να συμβάλλουμε στην οικοδόμηση μια ισχυρή οικονομική και ένωση και με την συμπερίληψη ενό backstop για τον ε, ε, μηχανισμού εξυγίανσης ε, και με άλλες μακροπροληπτικές ε, δράσεις. Και θα ήθελα να επισημάνω εδώ τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ESM του περασμένου Νοεμβρίου, που υιοθετήθηκε και από την Σύνοδο Κορυφής. Φιλοδοξία μα είναι η νέα συνθήκη να συμπεριλαμβάνει και δέσμευση ενσωμάτωση του ESM στο ενωσιακό πλαίσιο το σεμότερο δυνατόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο. Και τώρα. Έχουμε τώρα τους ομιλητές από τις διάφορες επιτροπές, αλλά δεν βλέπω εδώ τον Καταλήν Σορίν Ιβάν από την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Θα δώσω πάρα αυτά λοιπόν το λόγο στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, να ακούσουμε την άποψη της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. κυρία Χιούμπνερ έχει το λόγο. Έχετε ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Θεωρώ ότι κάποια θέματα είναι πολύ σημαντικά για την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων και είναι δύο αυτά τα σημαντικά θέματα που θα να θέσω. Καταρχά, τη συμπερίληψη του διαδόχου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητα στο νέο τάξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι λεπτομέρεια, είναι βασικό στατικό τη πρόταση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά επανάληψη ζητάει να σταματήσουν αυτέ τι διακυβερνητικέ ε, διευθετήσει που πριτάνεσαν κατά τη διάρκεια τη ε, κρίση και να ενσωματωθεί στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε μια καλή ευκαιρία. Επίση, τα κράτη-μέλη θέλουν να τροποποιήσουν τη συνθήκη ε, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητα, αλλά θα πρέπει να δούμε πολύ σύντομα το θέμα τη ενσωμάτωση στην ανομή τάξη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, ε, ο διάδοχο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητα είναι σημαντικό για το Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να έχουμε με ένα μηχανισμό, τόσο ώστε να υπάρχει λογοδοσία των αποφάσεων του διαδόχου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητα και η πρόσβαση τη πληροφορία είναι προπόθεση για να υπάρξει λογοδοσία. Θα πρέπει να υπάρχει υψηλό επίπεδο σε ό,τι αφορά τι αποφάσεις που παίρνει ο διάδοχο φορέα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητα, η διάδοχη κατάσταση. Ευχαριστώ την κυρία Χιούμπνερ. Και τώρα θα ακούσουμε τις πολιτικές ομάδες. Ξεκινάμε το ΕΛΚΑ. Ο κύριος Βάντεν Κέντερλε. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, συνάδελφοι. Η οικονομική κρίση μας έφερε αντιμέτωπους με την πραγματικότητα ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η Νομισματική Ένωση ε, και οι εθνικές ευρωπαϊκές αρχές κάπως ε, ήλεγχαν ε, τις εθνικές τράπεζες αλλά δεν είχαν καμία εικόνα της συστημικής κρίσης και καταστροφής που ερχόταν κατά πάνω μας. Και κάποιοι τελικά χρειάστηκαν, χρειάστηκε να διασωθούν από την Ευρώπη. Δημιουργήθηκε λοιπόν ο ESM και έκανε ξεκάθαρα αυτό που όφιλε να κάνει. Είναι σημαντικό όμως να τονίσουμε εδώ ότι ο Ευρωπαϊκό Μηχανισμός Διάσωσης πάντα ε, παραμένει ένας μηχανισμός έκτακτης ανάγκης. Θα πρέπει ε, όποιος ε, βρίσκεται σε κατεπίγουσα ανάγκη να έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί σε ένα τέτοιο μηχανισμό. Να υπάρχουν όμως ε, επαρκή αποθέματα οικονομικά ε, για τις στιγμές που πραγματικά θα χρειαστούν. Και εξάντε λοιπόν έχουμε προϋποθέσεις και εξ να προσαρμόζουμε στην ε, πραγματικότητα δεν πρέπει να αποδυναμώσουμε την πρόταση, γιατί, ε, να αποδυναμώσουμε τη δημοσιονομική πειθαρχία, γιατί ξέρουμε ότι η Ευρώπη έτσι κι αλλιώ θα έρθει να σώσει όποιον χρειάζεται βοήθεια. Δεν θα θέλατε, κύριε Πίτροπε, να σας ε, καλέσουμε μια ωραία πρωία χωρίς καμία προϋπόθεση. Πρέπει λοιπόν να τεθεί επικεφαλή ε, του θεματολογίου αυτό το ζήτημα, μαζί και με την ε, ενίσχυση ε, τη κεφαλοαγοράς στην Ευρώπη. Νομίζω ότι είναι ένα απαραίτητο βήμα λοιπόν για να καταστήσουμε πιο ανθεκτική την Ευρωζώνη επέναντι σε κρίση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, συγγνώμη. Τώρα η κυρία Περδόν Μπερές από τους Σοσιαλιστές για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαιρόμαστε που έχουμε την ευκαιρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο να εκφράσει την απόψη του για το πώς θα εξελιχθεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας με αυτή την ενδιάμεση έκθεση. Προφανώς αυτή η συζήτηση μπλοκάρεται 100% στο Συμβούλιο. Η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ήταν μια επιτυχία τη στιγμή που κάποια κράτη-μέλη χρειαζόντουσαν κάτι τέτοιο για να διασωθούν και δεν είχαν πια πρόσβαση στι αγορέ. Αυτή η επιτυχία σήμερα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να περάσουμε σε μια νέα φάση. Και ξέρουμε ότι αυτή η νέα φάση συνδέεται με ένα νέο πλαίσιο, όπου το θέμα του επιμερισμού των κινδύνων και της μείωσης των κινδύνων ε, έχει περάσει σε άλλα επίπεδα και με την υιοθέτηση του πακέτου για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και με το πακέτο ε, για τις τράπεζες. Γι' αυτό λοιπόν η ομάδα μου πιστεύει ότι η εξέλιξη αυτού του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητα δεν θα πρέπει να δημιουργήσει στην ε, δημιουργία ενό Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου. Θα θέλαμε πάρα πολύ να δημιουργήσουμε ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Σταθερότητα. Ε, η συμφωνία θα, αφορεί, θα αφορά το αν θα διατηρηθεί το ισχύον όνομα. Ε, ο μηχανισμό αυτό θα πρέπει όμω ε, να δούμε τι θα κάνει στο μέλλον. Για το μέλλον θα θέλαμε να χρησιμοποιείται πλήρως αυτό ο μηχανισμό για να εξασφαλίσει σταθερότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίω στην Ευρωζώνη ή να βοηθήσει αυτούς που έχουν ανάγκη να δώσει τις εγγύησεις που χρειαζόμαστε ε, στα πλαίσια του περίφημου backstop, του μηχανισμού ασφαλείας του τραπεζικού τομέα. Ξέρουμε ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίε. Υπάρχουν πάρα πολλά που εξελίσσονται στο Συμβούλιο. Φοβάμαι όμω ότι ε, αυτό ο μηχανισμό ε, σταθερότητα ε, είχε ένα λάτωμα στη γέννησή του και αυτό συνεχίζεται. Όταν τότε δεχτήκαμε να δημιουργηθεί αυτό ο μηχανισμό σε ένα διακυβερνητικό πλαίσιο ήταν γιατί είχαμε φοβερή ανάγκη. Υπήρχε κατεπίγουσα ανάγκη και θεωρούσαμε ότι θα διορθώσουμε αργότερα αυτή την κατάσταση. Σήμερα το Συμβούλιο όμως δεν θέλει να ακούσει τίποτα, καμία κουβέντα για τη χρήσιμη πρόταση που έκανε η Κομισιόν και έθεσε επιτάπητος, που θα μας επέτρεπε να προχωρήσουμε και να υπάρξει μια ενσωμάτωση αυτού του μηχανισμού στις συνθήκες. Και αυτό που θέλει το Κοινοβούλιο και ζητάει μετεπιτάσεως, ε, θεωρεί ότι είναι καλύτερη ε, οδός για το μέλλον αυτού του μηχανισμού. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε την κυρία Μπεχές. Και τώρα από το ECR, Ραρτ Πάκετ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με αυτή την έκθεση θέλουμε ουσιαστικά και τον ESM και τη δημοσιονομική αρρωγή προς τα κράτη-μέλη να τα ενσωματώσουμε άπαξ και διαπαντός στο ενωσιακό πλαίσιο. Και η δημοσιονομική αρρωγή εδώ θεωρείται ως βασικό μέλημα και καθήκον. Εμείς δεν συμφωνούμε. Το να δίνουμε περισσότερα χρήματα δεν λύνει κανένα πρόβλημα, γιατί τελικά το δημόσιο χρέο θα παραμένει πάντα δαμόκλειο σπάθη πάνω από τα κεφάλια των Ευρωπαίων πολιτών. Πρέπει να βρούμε άλλα κίνητρα και άλλε λύσει για να αναλάβουν ε, τα κράτη-μέλη τι ευθύνε του. Είναι λογικό λοιπόν να αφήσουμε την σχέση με τον ESM ε, στα κράτη-μέλη, γιατί εκείνοι διαχειρίζονται αυτά τα κονδύλια. Τα εθνικά κοινοβούλια είναι αυτά που θα αποφασίσουν. Εμείς δεν πρέπει να επικεντρωθούμε στις ε, νέες διασώσεις χωρών, αλλά στην πρόληψη κρίσεων. Και αυτό γίνεται ε, με τους δημοσιονομικούς κανόνες και την περαιτέρω εξέλιξή τους. Γιατί όταν μια χώρα δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τα χρέη τη, θα πρέπει να βρούμε άλλες λύσεις. Δεν γίνεται να επομίζεται ο ένας τα προβλήματα του άλλου. Και πρέπει να υπάρχει η ρήτρα και να επιστρέψει η ρήτρα του no bailout στην Ευρώπη, γιατί δεν ε, χρειάζεται εδώ να επανεφεύρουμε τον τροχό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Πάκετ. Από τους φιλελεύθερους, ο Δύο Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να χαιρετήσω την εξαιρετική εργασία που κάνουν οι δύο συνεισηγητέ. Και χαίρομαι όλου ιδιαίτερω που μπορούμε να μιλάμε για αυτό το νέο μηχανισμό χρηματοπιστωτική σταθερότητα στα πλαίσια του ενωσιακού δικαίου, τη ενωσιακή ενόμη τάξη. Όταν δημιουργήσαμε το ενίο νόμισμα, δεν μπορούσαμε να έχουμε φανταστεί τότε την οικονομική κρίση στην οποία θα βρισκόταν μετά από κάποια χρόνια η Ευρωζώνη, κυρίω λόγω τη κρίση δημοσίου χρέου και εξαιτία των δυσκολιών που γνώρισε η Ελλάδα. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό χρειάστηκε να δημιουργήσουμε ένα όργανο προκειμένου να καταφέρουμε να βοηθήσουμε ορισμένε χώρε με το πολύ υψηλό επίπεδο δημοσίου χρέους. Είναι πολύ σημαντικό μηχανισμό αυτό, ο ευρωπαϊκό μηχανισμό Σταθερότητα να ενταχθεί στην ένωμη τάξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και χαίρομαι όλου ιδιαίτερω που οι συνεισηγητέ είπαν ότι θα πρέπει να υπάρχει στενός δεσμός με τα εθνικά κοινοβούλια λέγοντα ότι θα πρέπει αυτό ο ευρωπαϊκό μηχανισμό χρηματοπιστωτική σταθερότητα να έχει μια έντονη κοινωνική πτυχή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν τα εθνικά κοινοβούλια να επιληφθούν επ' αυτού. Τα εθνικά κοινοβούλια είναι αυτά τα οποία αναλαμβάνουν ναι, τι δεσμεύσει σε εθνικό επίπεδο. Να πω όμω ότι λυπάμαι και για κάτι. Μιλάμε εδώ πέρα για την διακυβέρνηση τη Ευρωζώνη και λυπάμαι που δεν προβλέπεται εδώ πέρα ένα υπουργό οικονομικών, ένα αντιπρόεδρο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο οποίο θα μπορούσε να είναι αρμόδιο για την Ευρωζώνη. Θα ήθελα επίση να εκφράσω και μια επιθυμία, μια ευχή η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει το νόμισμά της όπως οι Ηνωμένε Πολιτείε προκειμένου να τηρηθούν σε διεθνές επίπεδο και σε εξωγραφικό επίπεδο οι βασικές αρχές και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω κάποια στιγμή στο μέλλον να καταφέρουμε να χρησιμοποιήσουμε το ευρώ ως αμυντικό μέσο προκειμένου να καταφέρουμε πραγματικά να προασπίσουμε τα ζωτικά μας συμφέροντα. Να ευχαριστήσω για άλλη μια ακόμα φορά τους δύο συνεισηγητές για την εξαιρετική τους εργασία στα πλαίσια αυτής της προσωρινής έκθεσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Αρτουή. Ο κύριος Σουρτάσουν τώρα, εξ ονόματος των Πρασίνων. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι η πρόθεση πίσω από τον μηχανισμό χρηματοπιστωτικής σταθερότητας ε, ε, είναι καλή. Δυστυχώς δεν κάνουμε αυτό ακριβώς. Αυτό που κάνουμε είναι ότι θεσπίζουμε ένα μηχανισμό που θα εξακολουθεί στην πράξη να είναι ενδο, ενδο, ε, σε ένα κοινοτικό κεκτημένο. Επίσης έχουμε πρόβλημα με το ρόλο του Κοινοβουλίου σε αυτή τη μεταρρύθμιση. Το είπαν και κάποιοι συνάδελφοι. Θα έπρεπε να είμαστε στη διαδικασία της συναπόφασης, όχι της συγκατάθεσης, όπως υποχρεωνόμαστε. ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός, ε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ε, είχε, έπαιξε σημαντικό